δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έχετε το λόγο κυρία Μογκερίνη. Uh, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να αρχίσω αναφερόμενοι στο άρθρο 36 που λέει ότι είπα το εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις κύριες πτυχές και επιλογές της κοινή πολιτικής ε, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και για την εξέλιξή τους. Στη συνέχεια λέει αυτός ή αυτή προφανώς θα λαμβάνει υπόψη τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω λοιπόν ότι τον τελευταίο χρόνο καταφέραμε επιτυχώς να υλοποιήσουμε τόσο αναφέρει αυτό το άρθρο. Είχαμε διαβουλεύσεις τακτικά εδώ, ενημερώσεις, ακούσαμε τα σχολιά σας, είχαμε συνεχή διάλογο για την εξωτερική μας πολιτική. Όμως, επιτρέψτε μου Πρόεδρε επίσης να πω ότι έχοντας πέντε συζητήσεις έχουμε δύο ώρες καθυστέρηση, κάτι το οποίο δεν είναι καλό ούτε για εσάς ούτε για μένα. Η καθυστέρηση αυτή με την οποία αρχίζουμε τη σημερινή συζήτηση. Κατόπιν τούτου πρέπει να σας πω ότι η φετινή χρονιά ήταν πολύ απαιτητική όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Η ευρωπαϊκή διπλωματία, κυρίως για το θέμα της Συρίας, δούλεψε πολύ. Και οι χώρες μέλη για πρώτη φορά ενεργοποίησαν το άρθρο 42-7 κάτι το οποίο αποφασίστηκε εδώ στο επικύκλιο αυτό. Όσον αφορά τώρα το προσφυγικό, επίσης συζητήσαμε και ενεργοποίησαμε πάρα πολλά εργαλεία. Το Σοφία, στο κέντρο της Αφρικής επίσης, ε, την βοήθειά μας στους καταβλισμούς για προσφύγους, στο Λίβανο, την Τουρκία. Όλα αυτά μαζί τα υλοποίησαμε. Οι προκλήσεις ήταν πολλές η εξωτερική πολιτική στρέφεται πολλές φορές και στις Ηνωμένε Πολιτείε βρίσκεται σε προεκλογική εκστρατεία, δεν είναι ε, μια χρονιά όμως κατά διάρκεια της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει ρεπό, κάθε άλλο. Η αδράνεια μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να επιδεινώσει τα πράγματα. Στη συζήτηση αυτή θα αναφερθώ στις άμεσες προτεραιότητες της εξωτερικής μας πολιτικής και αν έχουμε περισσότερο χρόνο για το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο όσον αφορά την στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην εξωτερική πολιτική, αυτό θα το κάνουμε αργότερα. Δεν βλέπω κανένα λόγο να έχουμε δύο συζητήσει για θέματα τα οποία είναι παρόμοια μεταξύ του και αυτό μέσα στην ίδια ημέρα. Α εξοδεύουμε το χρόνο μα πιο αποτελεσματικά και πιο λογικά. Λοιπόν, έρχομαι στι προτεραιότητέ μα. Πρέπει να σταματήσει ο εμφύλιο πόλεμο στην Μέση Ανατολή και την Αφρική. Αυτό είναι η πρώτη μα προτεραιότητα. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος γίνεται σε διαφορετικά μέτωπα ανάμεσα στη Συρία, το Ιράκ και την Τουρκία αλλά και στην Ιαμένη και την Λιβύη. Το κάθε μέτωπο έχει τη δικιά του ιστορία και τους δικούς του πρωταγωνιστές και τη δικιά του εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση όμως η λύση στη σύγκρουση πρέπει να έρθει μέσω της εθνικής συμφιλίωσης. Τας, αλκαΐδα και άλλες τρομοκρατικές ομάδες ε, δεν μπορεί να περάσουμε μέσα από αυτή την πολιτική διαδικασία. Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Παγίωση των ε, δυνάμεων επιτόπου που θα σταματήσουν τον πόλεμο. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη συμφιλίωση και να δουλέψουμε για κάποιο είδους ειρήνη. Στη Συρία κάτι πάει να γίνει, κάτι που φαινόταν απίθανο πριν από μερικούς μήνες. Η κατάπαυση πυρός είναι βέβαια πολύ εύθραυστη, αλλά συνεχίζεται. Η ανθρωπιστική βοήθεια έχει φτάσει σε διάφορους θύλακες όπου βρίσκονται υπό πολιορκία. Μοστού και αλλού αρχίζει να στηρίζεται η διαδικασία συνομιλιών. Ήμουνα τον προηγούμενο μήνα στην Γενέβη και συναντήθηκα τους συμμετέχοντες στις συζητήσεις και συντονίζουμε με το G7 την θέση μας χτες τελευταία φορά. Χρειάζεται πρόοδος και χρειάζεται πολύ γρήγορα. Η ειρήνη έχει πολλούς εχθρούς και γι' αυτό επίγει το ζήτημα. Και εμείς πρέπει να βιαστούμε. Συγχρόνω χρειαζόμαστε και υπομονή, την υπομονή που μας έφερε εδώ. Οι διαπραγματεύσει δεν θα είναι εύκολες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και επίμονοι. Το ίδιο σκεί και για τη Λιβύη. Ε, περισσότεροι στο Ιντρίπολη συζητούν μετά από μήνες σκληρής δουλειάς προκειμένου υπάρξει μια έστω εύθραυστη συνένεση. Είμαστε στο σημείο κίνησης. Όλοι οι φορείς πρέπει να βοηθήσουν για τη μετάβαση εξουσία στη νέα κυβέρνηση. Και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο εκεί. Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής επ' αυτού όπως είμαι πάντα. Ό,τι και να κάνουμε θα το κάνουμε μαζί με τους Λίβιους. Αν ζητήσουν τη στήριξή μας θα τους δώσουμε τη στήριξη που χρειάζονται και επιθυμούν ανθρωπιστική βοήθεια, ε, κατάρτιση των δυνάμεων ασφαλείας, στο δικαστικό τομέα, τον έλεγχο των συνόρων. Το μέλλον όμως της χώρας είναι στα δικά τους χέρια. Η σταθερότητα της Λιβύης, η ευημερία της και η ήττα του Ντάς είναι θέμα εθνικής ενότητας. Η λύση της σύγκρουσης στη Λιβύη δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική και μόνο της Λιβύης. Η δικιά μας ευθύνη είναι να στηρίζουμε τη χώρα με συνέπεια. Τρίτον, για την περιοχή, η Εμένη. Τους επόμενους μήνες θα επικεντρωθούμε βέβαια στη Συρία και τη Λιβύη, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε και τα μάτια μας σε μια άλλη κρίση, ακόμα και αν αυτή δεν βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα. Η σύγκρουση στην Ιεμένη έχει οδηγήσει στην ανθρωπιστική κρίση μεγάλης κλίμακας. 80% του πληθυσμού τώρα χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια. Η αστάθεια επιτρέπει να ανθίζουν οι τρομοκρατικές ε, Ομάδε και στο κέρας της Αφρικής και στον Ειδικό ωκεανό και στη Μεσόγειο. Συναντήθηκα με τον ειδικό αποστολμένο του ΙΕ την προηγούμενη εβδομάδα και συνεργαζόμαστε για την κατάπαυση πυρό που άρχισε την Κυριακή που μα πέρασε. Συνοδεύουμε τη διαδικασία αυτή με συγκεκριμένη στήριξη, με την προετοιμασία διαπραγματεύσεων και έχοντα υπόψη μα την ευρύτερη περιοχή. Θα ολοκληρώσω αυτή την πρώτη προτεραιότητα με τη διαδικασία στη Μέση Ανατολή, γιατί παρά το γεγονό ότι δεν δίνουμε την ίδια σημασία δεν πρέπει να ξεχνάμε την Ισραηλινοπαστηλιανική διένεξη. Η επόμενη κλιμάκωση θα έρθει σύντομα αν δεν κάνουμε τίποτα. Μαζί λοιπόν με το υπόλοιπο μέρος του καρτέτου και με όλους τους εταίρους μας συνεργαζόμαστε για έκθεση με συστάσεις ουσιαστικές προκειμένου να βγούμε από το αδιέξοδο και να πετύχουμε τη λύση των δύο κρατών. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε και η δουλειά μας δεν έχει σταματήσει ποτέ. Μερικές φορές εργαζόμαστε ησύχως, αλλά πάντα όμως, πάντα εργαζόμαστε. Η κοινή γνώμη δεν επικεντρώνεται σε αυτό το πρόβλημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς σταματάμε το έργο μας. Πρέπει να τελειώσει η διανεξία αυτή και στη Λιβύη και στην Ιεμένη και στη Συρία αλλά και στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να υπάρξουν ισχυρές εταιρικές σχέσεις με τους γειτονές μας, αλλά και με τους κύριους παράγοντες στην Αφρική και την Ασία. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε την απειλή της τρομοκρατία, στην περιοχή, στον κόσμο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κλείσει το χάσμα το οποίο εκμεταλλεύεται η ΔΑΣ πρέπει να αποφύγουμε τη ζωσπαστικοποίηση και αυτό πρέπει να το κάνουμε με συμμαχία με τις περισσότερες μουσουλμανικές χώρες. Μόνο έτσι θα ενισχυθεί η ασφάλεια στην Ευρώπη, αλλά θα βελτιωθεί και θα ενισχυθεί και η ασφάλεια των εταίρων μας στη Μέση Ανατολή, στην ε, Βόρεια Αφρική, στην ε, ε, Ασία, στα Δυτικά Βαλκάνια. Το δεύτερο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και έχει να κάνει δεν είναι σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αλλά και εκεί η μετανάστευση και προσφυγικό συνεχίζεται, ακόμα και αν έχουμε ειρήνη στη Συρία. Μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών είναι μια πραγματικότητα πια και είναι κάτι που έχουμε συζητήσει και πρόσφατα εδώ. Η, ειρήνη δεν θα σταματήσει τις μετακινήσεις αυτές. Φυσικά ο πόλεμος επιδεινώνει την κατάσταση, δημιουργεί νέα κίνητρα ακόμα και για τους λαθροδιακινητές. Έτσι λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε με τους γειτονές μας να μην τους βλέπουμε σαν αντιπάλους ήμουνα στην Ορδανία και στην Αφρική πρόσφατα και παρατήρησα τα σκάφη της δικιάς μας επιχείρησης Σοφίας που έσωσαν εκατοντάδες ζωές το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Τρίτος τομέας όπου πρέπει επιγόντως να δραστηριοποιηθούμε είναι κάτι αυτονόητο αν θέλουμε να πετύχουμε τις άλλες μας προτεραιότητες και αυτό είναι οι πολυμερείς σχέσεις. Μόνο έτσι μπορούμε να λύσουμε τα παγκόσμια προβλήματα. Μπορεί να ακούγεται λιγότερο επίγον αν δεν λάβετε υπόψη σα σε τι ακριβώ μπορεί να βοηθήσει αυτή η πολυμερής διπλωματία. Και στο COP21 βοήθησε αυτή και σε άλλες συνομιλίες. Η πολυμερή διπλωματία κατέστησε εφικτή τη συμφωνία μας με το Ιράν. Αν υπάρχει μια συνολική προσέγγιση, λύση από την οποία έχουν να κερδίσουν όλοι, το καλύτερο σενάριο, αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο για την ευρωπαϊκή πολιτική. Και τη χρειαζόμαστε περισσότερο του επόμενου μήνε στον τομέα της μη διάδοσης. Η διεθνή κοινότητα έδειξε να συμφωνεί στο ζήτημα της Βόρειας Κορέας και έχουμε νέες εξελίξεις και στην Ουάσιγκτον συστήσαμε με τον πρόεδρο Ομπάμα αλλά και χτες ακόμα και με το G7 στην Χειροσύμα στην φλιβερή επέτειο που είχαμε. Είναι προς το συμφέρον όλων μας να συνεργαστούμε σε διεθνές επίπεδο για το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας και μης διάδοσης των πυρηνικών όπλων και του αφοπλισμού. Θα ολοκληρώσω για το ότι η πολυμερής συνεργασία θα μας βοηθήσει και στις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Στις περισσότερες συγκρούσεις, οποίες αναφέρθηκα μέχρι τώρα, είτε πρόκειται για το Ιράν, είτε τη Λιβύη, είτε Πακιστάν, είτε τη Συρία μερικώς, η ρωσική ηγεσία έδειξε να θέλει να συνεργαστεί με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Και αποφασίσαμε μαζί λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Υπουργούς δηλαδή πριν από μερικές εβδομάδες ότι θα συνεργαστούμε με τη Ρωσία εκεί όπου εμείς έχουμε συμφέρον να το κάνουμε. Ανακοινώθηκε και σήμερα επιβεβαιώθηκε νομίζω με τη σημερινή συζήτηση ότι θα υπάρχει νέα συνάντηση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ Ρωσίας μετά από πολλούς μήνες που δεν έγινε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα είναι κανονικές πια οι σχέσεις μας με τη Ρωσία. Ε, πιστεύω ότι ο κύριος Στόντεμπερκ ε, απάντησε με τα σωστά λόγια μια άλλη φορά όταν ερωτήθηκε ότι δεν θα επιστρέψουμε στο business as usual παρά μόνο εάν η Ρωσία σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Αυτά είπε. Η ευρωπαϊκή θέση υιοθετήθηκε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων πριν από ένα μήνα. Όλοι συμφωνήσαμε για πέντε αρχές της πολιτικής μας απέναντι στη Ρωσία. Επιλεκτική συνεργασία, σχέσεις με τους ανατολικούς εταίρους μας, ενίσχυση της αντοχής μας και στήριξη στην κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία. Όλα αυτά τα είπα πριν από ένα μήνα και επιτρέψτε μου επίσης να σας πω ότι όλες οι χώρες μέλη τώρα βρίσκονται στο ίδιο στάδιο. Και για τη Ρωσία αλλά και για τα περισσότερα άλλα θέματα. Απαιτείται η ενότητα αυτή έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τους δύσκολους αυτούς καιρούς. Νομίζω ότι σε όλα τα θέματα τα οποία ανάφερα πριν έχουμε κοινά συμφέροντα όλοι οι Ευρωπαίοι. Ε, οι πολίτες το γνωρίζουν αυτό, πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και οι κυβερνήσεις. Πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστικά κοινή εξωτερική πολιτική, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε καμία εξωτερική πολιτική. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τα μέσα και να αποκτήσουμε το βάρος το οποίο απαιτείται στην παγκόσμια σκηνή. Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν που μπορούμε να δώσουμε και υπολογίζω στην δική σας υποστήριξη για να διαμορφώσουμε την πολιτική ασφάλειας που απαιτείται στο μέλλον. Στο Μπρόκ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας είπατε. Με πολλά από τα οποία συμφωνώ. Ε, ήθελα όμως μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Βρυξέλλες να πω πως πρέπει να περάσουμε σε ένα νέο ορισμό της πολιτικής ασφαλείας. Δεν είναι πλέον τα κλασικά πράγματα. Το Ισλαμικό κράτος κάνει πόλεμο σε Συρία και ε, και Ιράκ κάνει οικονομικό πόλεμο στη Βόρεια Αφρική για να τσακίσει τον τουρισμό και έτσι βεβαίως από τους άνεργους να στρατολογήσει και τρομοκράτη στην Ευρώπη. Όλα αυτά γίνονται ταυτόχρονα και ταυτόχρονα και ενιαία πρέπει να είναι και ταυτόχρονα πρέπει να το δούμε και ενιαία πρέπει να είναι η απάντησή μας. Να δούμε δηλαδή τι θέματα και εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής αναπτυξιακής. περνάμε τα πράγματα διαφορετικά από του παρελθόν. Και βεβαίω εδώ πέρα πάει και η ενίσχυση της πολιτικής γειτονίας και η συνεργασία για την ειρήνη, την οποία αναφέρατε σε Συρία και Ιράκ, αλλά και στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε στο πλευρό εκείνων που θέλουν να δημιουργήσουν ειρήνη και πρέπει να ξεσκίσουμε κάθε επιρροή που ε, έχουμε. Και αυτό σχετίζεται και με τη μετανάστευση. Που και αυτήν πρέπει να τα δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής ειρήνης και ασφαλείας. Συνάδελφοι, πρέπει επίσης να πούμε ότι στο αποφασιστικό ζήτημα της κατάπαυσης του πυρός στην Συρία βλέπουμε πως οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι έδρασαν μόνοι τους και αναρωτιέμαι ότι μιλάμε συχνά για soft power, για το 60% της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας που το δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Αλλά όσο επιτυχής και αν είναι, είναι ακόμη πιο επιτυχής όταν υπάρχει και hard power από πίσω να τη στηρίζει. Το πρέπει λοιπόν να δούμε μέσω της συνθήκης Λισαβόνας πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια ενισχυμένη πολιτική άμυνας και ασφάλειας για να μπορούμε να κινούμαστε ε, με μεγαλύτερη στιβαρότητα. Αλλιώ πετάμε λεφτά. Και τέλος, κυρία Μογκερίνη, αναφερθήκατε στο θέμα της πολυμερούς διπλωματίας. Συμφωνώ. Πρέπει όμως σοβαρά κάποτε να μιλήσουμε για τον ποιο ρόλο παίζει η Ευρώπη σε έναν πολυπολικό κόσμο. Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε κάποιους δικούς μας ορισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλέκενστάιν. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, κύριε Μπροκ. Ο χρόνος σας δεν τελείωσε. Δεν πειράζει. Περισσότερος χρόνος για μένα. Ήθελα όμως να σας πω ότι έχετε δίκιο. Και βλέπει κανείς πως αλλάζει το περιβάλλον ασφαλείας. Πέρα από τις περιφερειακές συγκρούσεις στη γειτονιά μας έχουμε απειλές που δεν περιορίζονται γεωγραφικά απειλές όπως η τρομοκρατία, ε, το κυβερνοέγκλημα που πλέον δεν γνωρίζουν το όριο μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν στον τομέα των εξοπλισμών θα πρέπει να συνεργαστεί. Αν κάναμε κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να αποφύγουμε άλλη επικαλύψεις. Χρειάζεται λοιπόν συντονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας. Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως περισσότερους εξοπλισμούς, σημαίνει εξυπνότερη πολιτική προμηθειών. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση κινηθεί στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων και της πρόληψης κρίσεων για να είναι αυτόνομη θα πρέπει να έχει μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, γιατί η πολιτική ασφάλειας και η διπλωματία πάνε χέρι-χέρι. Μόνο όταν είναι και τα δύο επιτυχή μπορούμε να επιβάλλουμε τα συμφέροντά μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Φανόρντεν. θα περιοριστώ στα θέματα της ΚΕΠΑ. Εκ των προτέρων θα πρέπει να πω ότι η ομάδα των συντηρητικών δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο ΝΑΤΟ και στην βορειοατλαντική διάσταση γενικότερα. Είναι η ιδρυτική μας αρχή θα έλεγα. Δεν μπορεί να αναλάβει βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα προβλήματα του κόσμου ελαχιστοποιώντας τις προσπάθειες των άλλων. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει τις στρατιωτικές δυνατότητες πέραν του ΝΑΤΟ η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει κανένας λόγος για να εμπλακεί στρατιωτικά. Είναι μια πλήρη στρέβλωση το να θεωρήσει κανείς ότι η ΚΕΠΑ θα ενισχύσει το ΝΑΤΟ. Μπορεί να συμπληρώσει το ΝΑΤΟ μέσω ε, μη στρατιωτικών δυνατοτήτων. Αλλά αυτό αναιρεί τις ίδιες ε, τις αρχές της ΚΕΠΑ δεν μπορεί να δημιουργήσει στρατιωτικές αυτόνομες καταστάσεις στις οποίες δεν εμπλέκονται οι Ηνωμένε Πολιτείε, αν και πρέπει φυσικά να είναι, υπάρχει μια αιμονή με την ΚΕΠΑ, είναι κάτι το οποίο ε, απομακρύνει την προσοχή μας από τη σημασία του ΝΑΤΟ στην φάση κατά την οποία οι Ηνωμένε Πολιτείε δίνουν ανανεωμένη σημασία και βάρος. Μόνο Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες καταπολεμούν το ΝΤΑΕΣ γιατί φαίνεται ότι το ΝΤΑΕΣ είναι ο πιο άμεσος κίνδυνος στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στην ευμάρειά μας. Αντί λοιπόν να επενδύουν σε αμυντικές δαπάνες και να επιδεικνύουν πολιτική βούληση, στην ουσία χρησιμοποιούν ε, τις δυνατότητες τις οποίες παρέχει το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος της ομάδας των φιλελευθέρων θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρότασή σας, τις προτάσεις σας μάλλον, η Ευρώπη θα βρίσκονταν σε δυσκολότερη κατάσταση αν δεν υπήρχε η κοινή ε, εξωτερική πολιτική. Βέβαια είναι μια πολιτική η οποία δεν είναι και πάρα πολύ κοινή. 90 δις δίδονται ε, για την άμυνα της Ευρώπης και μόνο τα 5 δις προέρχονται από κοινέ επενδύσεις ενώ το 70% πηγαίνει σε κοινέ αποστολές. Ένα πολύ μικρό ποσοστό δηλαδή των κοινών δαπανών ε, καλύπτει τα θέματα της άμυνας. Αυτό είναι θα έλεγα η αδυναμία της ΚΕΠΑ. Ε, δεν έχει τα μέσα τα οποία απαιτούνται για να παρεμβαίνει αποτελεσματικά σε στιγμές κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ισχυρές χώρες στο εσωτερικό του Συμβουλίου Ασφαλείας των ε, Ηνωμένων Εθνών ε, δεν ε, κρίνουν πάντα με διαφορετικό τρόπο τα συμφέροντά τους σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να παρεμβαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να ελπίσουμε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αιστείες πολέμου στην Δυτική Ασία όπως επίσης και στο Βόρειο Αφρική να σβήσουν, να αντιμετωπιστούν για να καταλήξουμε σε μια επιτυχή παρέμβαση της Ένωσης. Η κυρία Λέζινγκ, το θέμα της δίκαιης κατανομής και εντός χωρών και μεταξύ χωρών είναι το σημαντικότερο θέμα όταν μιλάμε για την ειρήνη και την ασφάλεια. Το 2004 θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα δακτύλιο φίλων και καταλήξαμε σε ένα δακτύλιο φωτιάς γύρω-γύρω. Αξιολόγηση να γίνει σήμερα. Ε, είναι λίγο αργά. Και αν δεν τα καταφέρουμε δεν πειράζει περισσότερα λεφτά για όπλα. Δεν συζητάμε για την επίδραση της επιθετικής οικονομικής πολιτικής της Ένωσης που οδηγεί παραδείγματος χάρη σε καταστροφικές, ε, καταστροφικές συνέπειες οι εξαγωγές ε, βεβαίως ε, όπλων ε, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορειοαφρικής είναι θέμα αλλά δεν τις εμποδίζει τίποτα οπότε θα πρέπει να υπάρξει ακούμε ως πρώτο στόχος τα δικά μας τα συμφέροντα και κάπου μας ενοχλεί η δημοκρατία τα δημοψηφίσματα στην Ολλανδία για να κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα με στρατιωτικές παρεμβάσεις πάντα στο όνομα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μετά αυξάνεται πάλι η ανισότητα και γίνεται ακόμη πιο τεταμένη η κατάσταση και ούτω καθεξής. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, τώρα θα έχουμε και την χρήση κονδυλίων για στρατιωτικούς σκοπούς. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Υπάρχουν διάφοροι τομείς στους οποίους ε, οι πράσινοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα. Η πρόληψη μακροπρόθεσμα των συγκρούσεων, για παράδειγμα. Και εδώ πέρα δεν πρόκειται μόνο για την διπλωματία. Αυτό που εννοώ είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, τη φτώχεια, τις εμπορικές αθέμητες πρακτικές και υπάρχει βέβαια και αναπτυξιακή πολιτική που πρέπει να ενισχύσουμε. Κάποια παραδείγματα είναι αυτά μόνο για να έχουμε ένα καλύτερο κόσμο. Επίσης πρέπει να φροντίσουμε για την ασφάλεια των ε, ατόμων αλλά και διάφορες παραμέτρους Οπότε ενθαρρύνω τις χώρες μέλη να κάνουν περισσότερες προσπάθειες και να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ υπέρ της ειρήνης. Πρέπει να σέβονται όλες οι χώρες το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες κοινέ αξίες. Η συμφωνία με την Τουρκία, για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι είναι στο ύψος ε, των ε, αρχών αυτών που αναφέρω. Η Επίτροπος αναφέρθηκε στον αφοπλισμό. Ναι, είναι κάτι πολύ καλό. Πρέπει να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, να πετύχουμε τον αφοπλισμό αλλά να είμαστε πολύ προσεκτικοί και όταν εξάγουμε όπλα προς τρίτες χώρες. Η ασφάλεια είναι τελώς διαφορετική σήμερα στον κόσμο. Γίνονται διάφορες καταχρήσεις και οι φίλοι μας οι σημερινοί μπορεί να είναι εχθροί μας μεθαύριο. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τέτοιες πρακτικές και να αποφύγουμε και την ριζοσπαστικοποίηση των νέων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρβερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία της είπα της εκπροσώπου εδώ στο Μικύκλιο για να μας ενημερώσει και έτσι να μπορέσουμε και εμείς να ενημερώσουμε το εκλογικό μα σώμα πίσω στι περιφέρειές μα όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια και την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω πώ έχει οριμάσει μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα και ποιο θα είναι τα επόμενα βήματά μας δεν έχουμε πάντα αρκετές πληροφορίες για το κόσμο. Οι συναντήσεις γίνονται διακυβερνητικά ή απόρριτα. Σήμερα έχουμε μπροστά μας λοιπόν μία εκπρόσωπα η οποία θέλει να κάνει περισσότερα στην εξωτερική πολιτική και να υποστηρίξει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους χώρες, αλλά σαν μια συλλογική πολιτική. Είναι βέβαια υπεύθυνη για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την πολιτική μας άμυνα η ύπατος εκπρόσωπη αναθεωρεί τώρα την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια επαμβατική πολιτική και φάνηκε αυτό στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα δούμε όμως τι θα γίνει μετά το δημοψήφισμα τέλη Ιουνίου στη χώρα μου. Πρόεδρε, την προηγούμενη εβδομάδα δημοκρατικά οι Ολλανδοί απέρριψαν τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία. Και εγώ ενθαρρύνω τους Βρετανούς να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα και να απορρίψουν αυτό το σχέδιο που έχουμε μπροστά μας. Ας προστατεύσουμε τους εαυτούς μας από μια στενότερη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Μποργέζιο. Μας παρουσιάσατε ένα ιδηλιακό ε, θα έλεγα τοπίο. Ε, βέβαια υπάρχει εδώ ε, δυνατότητα να πούμε ότι έχουμε αποτύχει στον τομέα της ασφάλειας και μόνο προπαγανδιστικά μπορούμε να αναφερθούμε σε διάφορα θετικά σημεία και νίκες Βλέπω ότι θέλετε να υποστηρίξετε κοινότητες οι οποίες πανηγυρίζουν τη σφαγή των χριστιανών. Ε, τα πράγματα ε, έχουν αλλάξει. Δεν καταπολεμούμε αποτελεσματικά ε, τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Εσείς ενισχύετε την Αλνούσρα μόνο και μόνο γιατί είναι εναντίον του Σαντάτου. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε ότι η Τουρκία έχει δώσει τεράστιες ποσότητες όπλων προς οργανώσεις τέτοιου είδους και δεν λέτε τίποτα γι' αυτό. Και εύκολα ε, επίσης μπορείτε να δεχθείτε αλλαγές συνόρων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τον εξτρεμισμό που γεννά την τρομοκρατία και θα πρέπει να μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι οποίοι υπερασπίζονται την τρομοκρατία είναι τα τζαμιά που έχουμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Επιτίδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επί 15 περίπου χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά την αναγκαιότητα να υπάρξει κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Όμως, όσες εργατόρες και αν καταναλωθούν, όσοι τόνοι μελάνη και αν χυθούν δεν πρόκειται να υπάρξει κοινή εξωτερική πολιτική στην ευρωπαϊκή ένωση. ο λόγο είναι προφανή όσο η ευρωπαϊκή ένωση ήταν ένωση οικονομική τα συμφέροντα των κρατών μελών συνέπιπλαν ή εν πάση περιπτώσει υπήρχε η δυνατότητα να βρεθεί ένας τρόπος αυτά να συγκλίνουν. από τη στιγμή κατά την οποία η ευρωπαϊκή ένωση αποφάσισε να γίνει και ένα τρόπο των κρατών άρχισαν να γίνονται αντικρουόμενα. έχασε η ευρωπαϊκή ένωση τη συνοχή τη. η αλήθεια αυτή απεδείχθη πρόσφατα. προκειμένου να αντιμετωπίσουν το τσουνάμι αυτό των ε, προσφύγων και των παρανόμων μεταναστών πολλά κράτη έκλεισαν τα σύνορά του αδιαφορώντα εάν με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά καταργούσαν τη συνθήκη σέγγεν και το έκαναν αυτό διότι αυτό επέβαλε το συμφέρον του. Η Μεγάλη Βρετανία επισύει την απειλή του Brexit διότι αυτό επιβάλλει το συμφέρον τη. Ακόμη χειρότερα, η Γερμανία έχει κατορθώσει να κυριαρχήσει σε όλη την Ευρώπη με αποτέλεσμα να υπάρξουν κράτη τα οποία αντιδρούν επειδή θίγονται τα συμφέροντά του. Άρα λοιπόν, όση καλή θέληση και αν θέλουμε να επιδείξουμε, όση προσπάθεια και αν καταβάλουμε. Ευχαριστούμε, κύριο Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι θλιβερό που δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτά με την, τον κύριο, Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Υπόθηκε οι τρομοκρατικές επιθέσεις, ακόμα και αυτές πρόσφατα στις Βρυξέλλες, μας αναγκάζουν να αναρωτηθούμε για την αποτελεσματικότητα της κοινή εξωτερικής μας πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Και όπως είπε και ο Έλμαν, υπάρχουν και εσωτερικές επιθέσεις και εξωτερικές επιθέσεις. Εξάλλου γι' αυτό σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε λύση στη Συρία και τη Λιβύη αφενός και από την άλλη θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία των αστυνομικών μας αρχών, να έχουμε κεντρικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, κάποιες μόνο προτάσεις που εξετάζουμε, γιατί φαίνεται ότι η εξωτερική μας πολιτική είναι συνδεδεμένη τελικά και με την τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, Ευχαριστώ την είπα το εκπρόσωπο. Τώρα που συζητάμε για τα θέματα αυτά έχει αλλάξει το πλαίσιο σε σχέση με το 2014 που είχαμε ξανασυζητήσει. Οι δυνατότητες ε, ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθονται υπό αμφισβήτηση. Όσον αφορά την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μία εκτενή συνεργασία για να υποστηρίξουμε και να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεισφορά λοιπόν όλων των χωρών μελών απαιτείται χωρίς να διαφοροποιούμε τις χώρες κατά πόσο συμμετέχουν στο Σέγγεν ή όχι. Απέναντι στην τρομοκρατική απειλή είναι ζωτική σημασία να καθορίσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και όλα αυτά πρέπει να καθορίζονται πολύ συγκεκριμένα και όχι υποκειμενικά. Επίσης, πρέπει να συμμετάσχουμε περισσότερο στην επίλυση των συγκρούσεων που έχουμε στη Μέση Ανατολή και αυτό μαζί με τις χώρες της περιοχής. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερη σταθερότητα, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με απειλές στην ασφάλειά μας όλο και περισσότερες. Η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ δεν είναι πια υπομφισβήτηση. Οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν κύματα βίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τον ΝΑΤΟ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φωτίγκα έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπατή Εκπρόσωπε προϋπόθεση για να ασκηθεί μια κοινή πολιτική είναι να έχουμε μια κοινή αντίληψη των προκλήσεων και της απειλής. Η κοινή αντίληψη των απειλών δεν υπάρχει, ειδικά όταν μιλάμε για την Ρωσία. Βλέπουμε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και δυστυχώς οφείλω να πω πως η δική σας η γλώσσα κυρία εκπρόσωπε όταν περιγράψατε αυτά τα γεγονότα έχει αλλάξει από την ε, προηγούμενη φορά και ε, υπάρχει μια τελείως ε, ρωσοκεντρική αντιμετώπιση δεν αναφέρατε την Ουκρανία ούτε μια φορά πρέπει να ξαναδούμε και να ξανασκεφτούμε σοβαρά τις απειλές που αντιμετωπίζουμε αλλά και τους λόγους για τους οποίους η Ολλανδία ε, εκφράστηκε έτσι. Μήπως είχε σχέση με τη Ρωσία. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μπιουτικόφερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Μογκερίνη, αγαπητοί συνάδελφοι, οι πολίτες αναμένουν να αναλάβει τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο δεν το κάνουμε, υποσκάπτουμε την ίδια μας την νομιμοποίηση. Θεωρώ επίσης πως θα πρέπει να εκτιμούμε ρεαλιστικά τον ρόλο μας στο πλαίσιο του πολυμερούς ε, πλαισίου ασφαλείας. Ε, ειδικά με βάση τα όπα είπε και ο κύριος Φανόρντεν και κάποια άλλοι συνάδελφοι. Θεωρώ λοιπόν πως ε, θα πρέπει να έχουμε και πολυμερή διπλωματία αλλά να ενισχύσουμε και τα πολυμερή θεσμικά όργανα και να μην ε, καταλήξουμε σε μια νέα πόλωση ε, που θέλουν κάποιες άλλες δυνάμεις. Εν ολίγης θα ήθελα να αναφέρω τρεις πτυχές που είναι σημαντικές στο πλαίσιο μιας πολυμερούς πολιτικής. Πρώτον, διαπιστώνω πως η διαδικασία της ε, Βαρκελόνης ε, ξεκινούσε με αφετηρία μια κοινή πολιτική για τη Μεσόγειο, αλλά βλέπω πως τώρα η Μεσόγειος θεωρείται κάτι το οποίο μας χωρίζει και μας προστατεύει. Δεύτερον, χρειαζόμαστε μια στρατηγική εταιρική σχέση, ειδικά με την υποσαχάρια Αφρική. Και τρίτον, θεωρώ ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία με τις χώρες Αζίαν και ελπίζω να έχουμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση και σβήνει το μικρόφωνο του κυρίου Μπιτικόφερ. Σας ευχαριστώ. Κύριος Αρνότ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεωρεί την πολιτική της, ε, την εξωτερική της πολιτική και πολλοί εκπλήσονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι έχει εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι για λόγους διαφάνειας θα πρέπει να υπογραμμίσουμε κάποια πράγματα που λέγονται εδώ. Πέρυσι, για παράδειγμα, ο κύριος Γιούνκερ έκανε έκκληση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού στρατού. Αλλά είπε, δεν θα είναι για να τον χρησιμοποιήσουμε αμέσως. Το Σεπτέμβριο η Άγγελα Μέρκελ είπε στον Ντέιβιτ Κάμερον ότι δεν πρόκειται να επιτύχει μεταρρυθμίσει τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός αν την αντίθεση του προς, μια, προς ένα ευρωπαϊκό στρατό και ο Ντέιβιτ Κάμερον σιώπησε, ίσως υποχώρησε ίσως ε, απλά επέστρεψε τις Βρεξέλλες και φέρνοντα μας τρία πράγματα που είχαμε ήδη και ένα που δεν θέλαμε Αναρωτιέμαι πόσοι στο Ηνωμένο Βασίλειο γνωρίζουν ότι υπάρχει ευρωπαϊκό σχέδιο άμυνα το οποίο επίκειται για τον Ιούνιο λίγο μετά το δημοψήφισμα το επόμενο βήμα το οποίο θα είναι ο Ευρωπαϊκός Στρατός αλλά αν γνώριζαν ότι βρισκόμαστε υπό την απειλή ε, της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Στρατού δεν νομίζω ότι θα διακινδύνευαν την παραμονή του ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα επέλεγαν να φύγουν στις 23 Ιουνίου Ευχαριστώ κύριο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με βάση τα άρθρα 24 και 21 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στόχοι της κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προαγωγή της δημοκρατίας, της ε, ανθρωπιάς και των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολλές φανφάρες συνήψε αυτή τη συμφωνία με την Τουρκία και ε, αυτοί οι οποίοι ε, θέλαν να διδάξουν τους άλλους αξίες αυτές αυτοί είναι χαρούμενοι που κάποιος άλλος αναλαμβάνει την προστασία των εξωτερικών συνόρων μόνο που διάλεξαν λάθος άνθρωπο ο Ερντογάν είναι δεσπότης, είναι τύρανος αγνοεί τις μειονότητες εξισλαμίζει όλο και περισσότερο την Τουρκία και κάνει και διεξάγει ε, φίλο πόλεμο κατά του λαού του αυτή είναι η πολιτική μας και οι πολίτες δεν μπορούν πλέον να ακούν αυτά τα έολα επιχειρήματα. Αντί λοιπόν να μετακυλίουμε την ευθύνη πρέπει μόνοι μας να περασπιστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εφαρμόσουμε μια πολιτική με σπονδυλική στήλη και όχι με το καρνέ των επιταγών. Ο κύριος Κόρβιν Μίκε. Ευχαριστώ. Συνεχίζω τα τελευταία σχόλια. Κανονικά οι αυτοκρατορίες έχουν, εφαρμόζουν τις πολιτικές τους μέσω του στρατού τους. Εμείς δεν ε, έχουμε δικό μας στρατό. Προσπαθούμε να εξαγοράσουμε άλλους πολιτικούς ε, και χώρες στην Τουρκία για παράδειγμα για να προστεριστεί την πολιτική μας. Είδαμε όμως ε, τι είπε το Ολλανδικό Δημοψήφισμα για την Ουκρανία για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ολόκληρη ομάδα τρομοκρατών στον κόσμο που προσπαθούν να συναγωνιστούν μεταξύ τους για να ποιος πρώτο ευνηδιάσει ε, την Ευρώπη, κυρία Μογκερίνη. Και εμείς δείχνουμε μεγάλη αδυναμία. Εσείς είστε, κυρία Μογκερίνη, η απειλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιτίας της αδυναμίας που δείχνετε. Θεωρώ γι' αυτό λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταστραφεί. Η ε, κυρία Καρνιέτε. Κυρία Αντιπρόεδρε, Χαιρετίζω τα τελευταία βήματα για μια στενότερη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, δηλαδή έμπρακτη συνεργασία μεταξύ Frontex και ΝΑΤΟ στο Αιγαίο Πέλαγος. Η στενότερη συνεργασία με το ΝΑΤΟ ε, θα πρέπει να αποσοβήσει και απειλές στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει επίσης η υβριδική ε, και προκλήσεις και απειλέ να αντιμετωπίσουμε χάρη σε αυτή τη σύσφυξη της συνεργασία. Σας ενθαρρύνω λοιπόν να εφαρμόσετε το σχετικό έγγραφο και στα θέματα στενότερης συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, αλλά και στα υπόλοιπα 21 σημεία του σχεδίου δράσης. Προσβλέπω λοιπόν και στην θέσπιση των απαραίτητων νομοθετικών και πολιτικών μέτρων και στην γρήγορη εφαρμογή του. Ευχαριστώ. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν δώσω το λόγο ήθελα να επισημάνω ότι η υπηρεσία μας είπε πως έχουμε μεγάλη καθυστέρηση οπότε δεν θα δεχτούμε πολλές ε, μπλε κάρτες αν τις δεχτούμε και το ίδιο με το Catch the Eye. Το λόγο έχει ο κ. Χάουιτ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε στη συζήτηση του τελευταίου χρόνου για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας πριν το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ισχυρό στην Ευρώπη και η Ευρώπη είναι ισχυρή στον κόσμο οι αποστολές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κέρας Αφρική ελέγχθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο ε, η Ευρώπη ηγήθηκε τη συμφωνία με το Ιράν η διασκέψη για τη Συρία ήταν επιτυχής επειδή κατάφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τα τρία δις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο, αλλά συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Όλοι ασκούμε μεγαλύτερη επιρροή και αν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Σύμφωνα με Βρετανούς ηθήνοντες, η χώρα μου θα είναι λιγότερο ασφαλής και όπως υπόθηκε σήμερα αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα σε ολόκληρη την παγκόσμια τάξη. Στο σύγχρονο κόσμο διάφοροι σύμμαχοι, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, η Κίνα, όλοι λένε ότι είναι προτιμότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει ε, εντό ε, τη το Ηνωμένο Βασίλειο. Πώ είπε η Μέρκελ, μόνο ο Πούτιν θα χαρεί αν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο. σε όλη την ιστορία από τους, Ναπολε... από τους πολέμους των Ναπολέοντα μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τις πολιτικές εξελίξεις στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου η ε, το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχε στην Ευρώπη για τη διασφάλιση της ειρήνης δεν νομίζω ότι οι Βρετανοί ευρωσκεπτικιστές γνωρίζουν καλύτερα από την Επιτροπή Νόμπελ που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η επιτυχιαστή ε, ειρηνευτική διαδικασία στην ιστορία και εμείς είμαστε υπέρ αυτή τη ειρήνη και εγώ θα ψηφίσω υπέρ στο δημοψήφισμα για να παραμείνουμε. Σας παρακαλώ ε, να, διατηρείτε το, να τηρείτε το χρόνο. Ένα λεπτό κύριο Γιούρακ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, τελευταία, οι αρχέ Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, μερικές φορές ε, ε, επιτίθεται σε χώρες που προσπαθούν να προστατεύσουν τη, τα συμφέροντά τους. Ε, τελευταία είχαμε, πρώτα τελευταία είχαμε την Ουγγαρία, τώρα τελευταία την Πολωνία που απλώς ήθελε να, να εφαρμόσει μια πιο αντικειμενική έρευνα για να διαλευκάνει το, ε, το θάνατο στο αεροπορικό ατύχημα του Προέδρου της ε, του Λεχ Κατσίνσκι. Ε, ενώ ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε συζήτηση για, την, για το σεβασμό του κράτους δικαίου, γιατί υποτίθεται υπήρχαν μορφές κατά της Πολωνία, αλλά τίποτα συγκεκριμένο δεν ακούσαμε. Και τίποτα δεν έχει γίνει από την κυρία Μαγκελίνη τα τελευταία δύο χρόνια ούτε για να μας βοηθήσει. Και τώρα ούτε ακούμε για αυτό το πρόβλημα. Φαίνεται ότι είναι εύκολο να μιλούμε για την ε, η Εμένη, τη Λιβύη, να προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα του υπόλοιπου κόσμου, αλλά καμία βοήθεια προς τις ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Μορβά για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη, θα ήθελα να μου εξηγήσετε με σαφήνεια και με στοιχεία πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ξένων μαχητών. Γιατί τόσοι ξένοι μαχητές φεύγουν από εμάς για να πολεμήσουν το πλευρό του Ισλαμικού κράτους και τι γίνεται ε, με την επιστροφή τους. Και μόνο το ταξίδι συνιστά αξιόπινη πράξη. Μόνο η στρατολόγηση στο ίσις αποτελεί εξώπινη πράξη. Γιατί δεν έχουμε στοιχειοθετήσει αυτή την ενέργεια ως έγκλημα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να τυποποιήσουμε ένα ιδιώνυμο έγκλημα με, στην περίπτωση που κάποιος πηγαίνει να συστρατευτεί με το Ισλαμικό κράτος και από τη στιγμή που δεν είναι ο άνθρωπος αυτός υπήκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να απελαθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Τι γνώμη έχετε κύριε Μαγκερίνη. Κύριε Μογκερίνη, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για το διάλογο που κάνετε με μας με το Κοινοβούλιο. Ε, και βιώνουμε το εξής. Ε, όταν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά ως Ευρωπαίοι. Η συμφωνία με το Ιράν και η κοινή στάση ε, με τη Ρωσία στο θέμα της Ουκρανίας είναι ένα θέμα που ήθελα να αναφέρω. Τώρα, ε, αν αποτύχει όμως η όλη διαδικασία με τη Συρία, ως Ευρωπαίοι θα θυγούμε πολύ περισσότερο από ό,τι οι ΗΠΑ και η Ρωσία, διότι θα έχουμε νέες μεταναστευτικές ροές και πολλά άλλα. Για να μας πάρουν όμως ε, σοβαρά πρέπει να είμαστε και σκληροί και ήπια δύναμη. Αν ως Ευρωπαϊκή Ένωση στρατιωτικά μπορούμε να λειτουργήσουμε μόνο μέσα στο χώρο του ΝΑΤΟ, ε, καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε εξαρτώμενοι από βέτο του Ερντογάν. Στη Λιβύη θα πρέπει να ανοίξουμε και να διατηρήσουμε όλες τις δυνατότητες και τη συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση, αλλά ε, επίσης ε, να στραφούμε κατά της Αλκάιντα και των διακινητών. Ελπίζω η παγκόσμια, η σφαιρική στρατηγική που θα παρουσιάσετε θα περιλαμβάνει και μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ο κύριος Πεσκού για 1,5 λεπτό. Εάν ε, η άμυνα ήταν σε εθνικά χέρια, τότε τα εργαλεία της διαχείρισης της κρίσης θα ήταν ακριβώς αυτά από το να μιλάμε για κοινή άμυνα. Κοινή άμυνα, αυτό το έχουμε αφήσει στο ΝΑΤΟ, διότι οι συνθήκες αναφέρουν σαφώς ε, με την βοήθεια του άρθρου 42.7 και του άρθρου 222. Σήμερα όμως ε, όταν ζητάμε από τους Ευρωπαίους ή Διακόπτει η πρόεδρος. Πιο αργά κύριε Πάσκου, λέει η πρόεδρος. Κοιτάξτε, αν μιλάω όμως πιο αργά δεν θα προλάβω να πω αυτά που θέλω. Ε, είναι πιθανό να γίνει αυτό. Συνεχίζει ο κύριος Πάσκου. Πολλοί φοβούνται για τη ζωή τους, ε, κυρίως αυτά που έχουν κάνει οι τρομοκράτες. Κατόπιν τούτου η κοινή εξωτερική πολιτική ε, απολαμβάνει μια νέα χρειά, η οποία τώρα επισκιάζει την παραδοσιακή εξωτερική διάσταση, ακόμα και αν επιτύχουμε περισσότερα. Όσον αφορά την εσωτερική μας ασφάλεια, δέστε λιγάκι τον αριθμό των φορέων και στρατηγικών, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για βελτίωση βελτίωση κυρίως όσον αφορά τη συνεργασία ανάμεσα στις εθνικές αρχές και τους φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και τις ε, διάφορες άλλες ε, διεθνείς οργανώσεις. Κυρίως ε, όταν αναπτύσσονται στρατιωτικές δυνάμεις όπως έγινε στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι αυτοί παίρνουν όμως διαταγές από διαφορετικούς διοικητές. Έτσι λοιπόν πέρα από το να βελτιωθεί η σχέση ανάμεσα στις διεθνείς αρχές και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αρχίσουμε να ενσωματώνουμε ε, το, ε, την εργαλειοθήκη, την ε, πολιτική με την στρατιωτική για να έχουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση. Θα ήταν πολύ πιο απλό να είχατε ζητήσει δύο λεπτά αντί για ένα μισή λεπτό. Ο κύριος Μιγιάν Μον για ένα λεπτό. Και ανάψτε το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Μαγκερίνη για την παρουσίαση με την έξαρση του, της τρομοκρατίας ε, του Ισλαμικού κράτους, με την αστάθεια στη Λιβύη, στην Ουκρανία, στη Συρία, στο Ιράκ, ε, την κατάσταση στο Σαχέλ, την πίεση στα σύνορά μας, πολυάριθμες προκλήσεις, παγκόσμιες απειλές. Όλα αυτά δείχνουν ότι μια κοινή εξωτερική πολιτική την οποία προσπαθείτε να εφαρμόσετε δεν είναι πια επιλογή, είναι αναγκαιότητα. Ε, εν τη ισχύς μαζί θα είμαστε πιο δυνατοί. Και γι' αυτό μια εξωτερική πολιτική δεν θα πρέπει να έχει μόνο μέσα, αλλά και δεδηλωμένη πολιτική βούληση από τα κράτη-μέλη. Και ένα άλλο γενικό σχόλιο. Οι χώρες της γειτονίας θα πρέπει να κτίσουν πρωταρχικό ρόλο στην εξωτερική μας πολιτική. Αλλά θα πρέπει να ξεχνούμε και τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί υπάρχει αλληλεξάρτηση. Τίποτα δεν είναι μακριά. Ο κόσμος είναι διασυνδεδεμένος. Ε, ελπίζω λοιπόν το έγγραφο που θα υποβάλλεται στο Συμβούλιο τον Ιούνιο, κυρία Μογκερίνη, για την ε, σφαιρική πολιτική εξωτερικής ασφάλειας, ε, εξωτερικής και πολιτικής και ασφάλειας, να περιέχει και ένα κεφάλαιο για την εμβάθυνση στην πολιτική της ασφάλειας και της άμυνας. Ευχαριστώ κύριο Χάν για ένα λεπτό. Κυρία Υπατή εκπρόσωπε, η απόφαση για κυρώσει κατά της Μιανμάρ παρά της δημοκρατικής, ε, υπέρ της δημοκρατικής μετάβασης ήταν σωστή, αλλά έκτοτε η κατάσταση των ε, Ράγκα και των χριστιανών στη Μιανμάρ δεν έχει βελτιωθεί. Έχουμε αποδείξεις ε, ότι μπορεί να πρόκειται μάλιστα για γενοκτονία. Πέρυσι εδώ είπατε ότι δεν υπάρχουν όρια μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών γεγονότων. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τις δράσεις μας συμφώνησα μαζί σας τότε και συμφωνώ μαζί σας σήμερα. Όσοι ε, ε, διέπραξαν τις ε, επιθέσεις στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες ριζοσπαστικοποιήθηκαν διότι ξεπέρασαν αυτά τα όρια πρέπει να είναι οι δράσεις μας ε, γνωστές για να υπερασπίσουμε τις αξίες μας. Σας παροτρύνω λοιπόν να επαναφέρετε στην ατζέντα την ε, υπόθεση της Μιανμάρ και αν δεν σημειωθεί πρόοδος μέσα στις επόμενες εβδομάδες με την, με την νέα κυβέρνηση θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επιβάλλουμε πολιτική κυρώσεων. Ευχαριστώ ο κύριος Ντανζό για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε εκπρόσωπε, είναι πολύ δύσκολη η δουλειά σας και θλίβομαι που βλέπω ότι το κοινοβούλιο αυτό δεν σας διευκολύνει με τις ε, ατελείωτες συνεδριάσεις. Ε, δύο λόγια γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, ένα λεπτό είναι λίγος χρόνος για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Η παγκόσμια στρατηγική, η καθολική στρατηγική είναι αναγκαία όπως πρόκειται να την ετοιμάσουμε αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε μια άλλη προτεραιότητα την υλοποίηση των ήδη υπαρξών στρατηγικών η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δικές σας ε, υπηρεσίες ε, έχουν πληγεί από το πολυάριθμες στρατηγικές. Ε, κάθε υπηρεσία έχει και μια στρατηγική. Τραγικό παράδειγμα, σήμερα χάσαμε έναν 19χρονο στρατιώτη ε, Γάλλο στο Μαλί και υπήρξαν και πολλοί τραυματίες. Έχουμε μια στρατηγική για το ΣΑΕΛ εδώ και 10 χρόνια για την ασφάλεια και την ανάπτυξη, αλλά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί επαρκώς. Οπότε σας παρακαλούμε ναι παγκόσμια στρατηγική αλλά χρειάζονται και αποτελέσματα, υλοποίηση, ευελιξία και προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακτήσει την επιρροή στον κόσμο αν ε, επιβεβαιώσει θέση της ως ε, δύναμη μπορεί να αποτρέψει, να προβλέψει και έτσι να αποκτήσει μια σημαντική θέση στο παγκόσμιο προσκήνιο. Θέλουμε μια νέα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια που να ανταποκρίνεται στι νέε προκλήσει και του κινδύνου. Είχαμε τη διάλυση τη Λιβύη, τον εμφύλιο στη Συρία, τι δράσει του ΤΑΕ, την τρομοκρατία, τη σύγκρουση στο Σαχέλ, στο κέρα Αφρική. Θα πρέπει να επομιστούμε τι ευθύνε μα. Δεν μπορούμε να τι μετακυλούμε σε άλλου ε, διεθνείς παράγοντες. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας που θα ε, συνδυάζεται με την εξωτερική πολιτική, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αναπτυξιακή πολιτική. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προληπτικής, αποτρεπτικής και κατασταλτικής ε, ενέργειας και να συνεργαστούμε με άλλους ε, παγκόσμιους παράγοντες όπως είναι η Αφρικανική Ένωση, και ο αραβικό σύνδεσμο. Σα ευχαριστώ. Μιλήσατε όμω με πολύ μεγάλη ταχύτητα, κυρία Σύσο. Ο κύριο Κούκαν, για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ. Και ευχαριστώ την είπατε εκπρόσωπο για την εισαγωγή και την παρουσίαση που μα έκανε. Σήμερα περισσότερο από ποτέ νιώθουμε πόσο αλληλένδετη είναι η εξωτερική πολιτική και η εσωτερική μα ασφάλεια. Δυστυχώ γίναμε ευάλωτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή την άποψη. Θα πρέπει να ξανακαθησυχάσουμε του πολίτε μα ότι είμαστε ικανοί να έχουμε αποτελεσματικές εξωτερικές, εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλειας και πολιτική άμυνας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις πολιτικές μας εκεί που έχουν μεγαλύτερη αξία και βαρύτητα, στην εξωτερική πολιτική, στην ασφάλεια και στις γειτονικές μας χώρες, νότια-ανατολικά και με τους ε, εταίρους μας στα Βαλκάνια γιατί αλλιώς θα έχουμε ε, έξαρση και νέων απειλών και προκλήσεων που θα φτάνουν στην Ευρώπη. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και να ιεραρχήσουμε σωστά τις προτεραιότητές μας. Οι εξωτερικές μας πολιτικές θα πρέπει να έχουν νόημα. Για παράδειγμα, αν διευρύνουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια και βοηθήσουμε τους εταίρους μας προς Ανατολάς, δεν θα πρέπει αυτό να μας οδηγήσει να γίνουμε πιο εξαρτημένοι από το ρωσικό φυσικό αέριο. Δεν βλέπω τον κύριο Λάινεν στην αίθουσα και δίνω το λόγο στον κύριο Μακάλιστερ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε από την είπατε εκπρόσωπο ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστιες απειλές ε, και διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο ότι είναι ρευστά τα όρια ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια. Ε, είναι απαραίτητο να υπάρχουν περισσότερα κοινά στοιχεία ανάμεσα στην εξωτερική και την εσωτερική πολιτική. Και θέλω να επισημάνω ότι η πλειοψηφία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο πλευρό μας γιατί πολλές δημοσκοπήσεις Επίσης καταδεικνύουν ότι οι άνθρωποι επιθυμούν περισσότερα κοινά στοιχεία στην εξωτερική και την εσωτερική πολιτική. Η στρατηγική μας που πρέπει να υποβληθεί μέχρι τον Ιούνιο ε, πρέπει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις ε, και πρέπει επίσης ε, να καθορίσει τα απαραίτητα, τις απαραίτητες ε, διεθνείς ε, συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προς αυτή την κατεύθυνση σας εύχομαι καλή επιτυχία κυρία Μογκερίνη. Πολύ ωραία, περνάμε τώρα ε, στη διαδικασία Catch the Eye. Για ένα λεπτό. Η κυρία Βιρκούνεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όλο και πιο δύσκολη. Η εξωτερική πολιτική είναι ελεύθερη με την εσωτερική ασφάλεια. Έχουμε τρομο, απειλή της τρομοκρατίας, μεταναστευτικές και προσφυγικές πιέσεις, θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε την προστασία και την ασφάλεια. Και ταυτόχρονα οι παραδοσιακές στρατικές απειλές δεν έχουν εξαφανιστεί. Απόδειξη η επιθετική στάση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Για τις χώρες της Ευρώπης το ΝΑΤΟ είναι μια στρατιωτική λύση. Δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτιάξει μια αντίπαλη δομή σε σχέση με τον ΝΑΤΟ. Απλώς θα πρέπει να ενισχύσουμε με τη συνεργασία μας τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ και θα πρέπει να αναλάβουμε περισσότερο τις ευθύνες της άμυνας στην Ευρώπη. Και αρχή της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας είναι η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κράτη-μέλη της. Δεν είδα όμως καμιά αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα κατά των παρανόμων ενεργειών των σκοπίων. στις 29 μαρτίου σας υπέβαλα γραπτή ερώτηση με προτεραιότητα με την οποία σας ζητούσα να λάβετε μέτρα κατά των σκοπίων διότι στα μέσα μαρτίου η αστυνομία των σκοπίων επιτέθηκε κατά προσφύγων που ήταν εντός του ελληνικού εδάφους στην ιδωμένη ρίχνοντας δακρυγόνα και χημικά. όμως δεν έγινε τίποτε και την προηγούμενη κυριακή αποθρασύνθηκαν τα σκόπια επετέθηκαν στους πρόσφυγες είχαμε πολύ περισσότερους τραυματίες πυροβόλησαν και έριξαν σφαίρες με καουτσούκ και είχαμε πάρα πολλούς τραυματίες. για ποιο λόγο λοιπόν γίνονται αυτά. εάν είχατε απαντήσει έγκαιρα την ερώτηση που σας είχα υποβάλει με προτεραιότητα εντός δέκα ημερών τότε ίσως στις 8 Απριλίου να είχατε απαντήσει και να είχατε κόψει το βήχα στους Σκοπιανούς. Περιμένω μια απάντηση έστω και τώρα. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε Μογκερίνη. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη ευκαιρία που είχαμε για ε, έντονο διάλογο με τους ευρωβουλευτές. Ε, αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ευκαιρία τέτοια συζήτησης. Ε, στις επιλογές εξωτερικής πολιτικής ε, και για να γίνουμε ε, παράγων που βαρύνει στην παγκόσμια σκηνή θα πρέπει να απαντήσουμε σε τρία ερωτήματα. Ε, καταρχήν, το θέμα της σύνδεσης εξωτερικής πολιτικής και εσωτερικής ασφάλειας μετά τις ε, τρομοκρατικές ε, απειλές και την ανάγκη να ελέγξουμε το προσφυγικό βήμα. Επίσης, σχέσεις με την Τουρκία. Εκεί έχουμε και αστάθεια στην περιοχή και μια ενταξιακή διαδικασία και τον έλεγχο της μετανάστευσης και την εποπτεία των εξωτερικών μας συνόρων. Και ένα τρίτο σημαντικό θέμα είναι η Ουκρανία είδαμε ότι στις κάτω χώρες ένα εθνικό δημοψήφισμα με ευρωπαϊκό θέμα έχει και διεθνείς συνέπειες. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τις, τις ε, συνέπειες που έχουν οι δραστηριότητες μας στην εξωτερική πολιτική και οι δραστηριότητες μας γενικώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε με το ΚΑΤΣΔΙ. Το λόγο έχετε και πάλι εσείς κυρία Μογκερίνη. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω και νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα πάτησα στην επιστολή σου, οπότε θα τη λάβετε μάλλον αύριο το πρωί, το έλεγξα με τους συνεργάτες μου. Θα ήθελα να τονίσω αυτά που είπαν πολλοί προλαλήσαντες ε, για το σχετισμό της ε, εξωτερικής ε, ασφάλειας με την εσωτερική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα στο Κοινοβούλιο συζητήσαμε δύο πτυχές της εσωτερικής πλευράς της ε, πολιτικής μας, που έχει όμως και εξωτερική διάσταση. Ε, πώς θα ανταποκριθούμε στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση και τι θα γίνει με την αντιτρομοκρατία. Πώς θα καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία μετά τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις της Βρυξέλλες. Οπότε οι πολιτικές μας έχουν και εσωτερική και εξωτερική πτυχή. Και τους τελευταίους μήνες μάλιστα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στο Συμβούλιο θετήσαμε μια προσέγγιση ώστε να έχουμε πιο ολοκληρωμένη ε, αντιμετώπιση των εσωτερικών και εξωτερικών πτυχών θα σας ενημερώσουμε ε, σύντομα για την ε, σφαιρική μας στρατηγική. Γιατί αυτό είναι το νόημα της ε, σφαιρικής στρατηγικής. Η συγχώνευση διαφόρων πτυχών πολιτικών που έχουμε στα κοινοτικά θεσμικά όργανα για να ξεπεράσουμε τα κενά που έχουμε σήμερα και τα χάσματα που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν για τη χρήση των εξωτερικών και εσωτερικών εργαλείων. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι η συζήτηση έδειξε ότι και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο θα πρέπει να αναπτύξουμε νέους τρόπους σκέψης και αντιμετώπισης των προκλήσεων. Γιατί όταν συζητούμε για τις εσωτερικέ πτυχές και την τρομοκρατία αλλά και τις εξωτερικές πτυχές ουσιαστικά σε δύο διαφορετικές συναντήσει, σε δύο διαφορετικέ συζητήσεις μιλούμε για τα ίδια θέματα. Οπότε θα πρέπει να βρούμε καινοτόμους διαφορετικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε το ίδιο θέμα υπό διαφορετικά πρίσματα και σκοπιές. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τόσο διαφορετικά εργαλεία, εξωτερικά, εσωτερικά, ήπια, σκληρά και μία γενικώ σφαιρική προσέγγιση. Αλλά μερικές φορές ε, εμεί είμαστε οι πρώτοι που ενώ πρεσβεύουμε την σφαιρική και περιεκτική προσέγγιση δεν την εφαρμόζουμε. Βέβαια πολλά σχόλια από αυτά που ακούσαμε εκφεύγουν τη σημερινή συζήτηση. Αναφέρθηκε ο ορισμός του ρόλου μας στον κόσμο. Ο κύριος ε, Μπρόκ χαρακτήρισε τον κόσμο ως πολυπολικό. Πολύ αμφιβάλλω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε πόλους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε πολυπολικό κόσμο, γιατί δεν βρίσκουμε τους πόλους. Έχουμε έναν ε, μεταβαλλόμενο συνεχώς κόσμο. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, άλλη συζήτηση. Ο κύριος Ντανζόν ε, μίλησε για κάτι κέριο, το πώς θα εφαρμόσουμε τις στρατηγικές που εκπονούμε και θεσπίζουμε. Θα ήθελα ε, το θέμα αυτό να το συζητήσουμε στα πλαίσια της παγκόσμιας στρατηγικής, γιατί η εφαρμογή είναι ουσιώδη στοιχείο της ε, στρατηγικής. Δεν είναι η συνέπεια το τέλος, αλλά είναι αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής μας. Ένα άλλο θέμα που επισημάνθηκε είναι ότι και πολλές άλλες πολιτικές και πολλές άλλες προτεραιότητες σε βασικούς τομείς τους οποίους δεν ανέφερα σήμερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή τους ανέφερα δεν είναι και προτεραιότητες. Εγώ αναφέρθηκα σε τρεις. Ενεργειακή ασφάλεια, αναφέρθηκε πριν από λίγο. Οι σχέσεις μας με τις χώρες ΑΣΕΑΝ, αναφέρθηκε από κάποιον προλαλήσαντα. Άρτη αφιχθής από την Ιαπωνία για το G7, ε, και στη Τζακάρτα, είχαμε εξαιρετική συνεδρίαση με τον γραμματέα της ΑΣΕΑΝ και τα κράτη-μέλη για, για το πώς θα αναβαθμίσουμε τις ε, σχέσεις μας και να τις κάνουμε στρατηγικές. Και επίσης Σαχέλ, κέριο θέμα για την ασφάλειά μας και για τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, αλλά ναι, ευρωπαϊκή σημασία θα έχει και για, την για τις οικονομικές εξελίξεις και για τα παγκόσμια ζητήματα. Πάντως, επαναλαμβάνω, προσπάθησα να επικεντρωθώ στις άμεσες ε, και πιο επιτακτικές προτεραιότητες που αντιμετωπίζουμε, που έχουμε. Τέλος, ε, να πω δύο λόγια για ένα θέμα που σχολιάσατε πολύ. Την προστιθέμενη ή μη προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Εγώ βλέπω στους συμπολίτες μας όλο και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ε, και στα κρατημέλη, ότι ούτε και τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη δεν είναι πια παγκόσμιες ε, δυνάμεις. Γιατί έχουμε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύο κατηγορίες χωρών, τις μικρές χώρες και αυτές που δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι μικρές. Αλλά αυτή, αυτό είναι το δείγμα της ιστορίας και αυτό αφορά την εξωτερική και την πολιτική ασφαλεία μας. Τίποτα ε, δεν μπορεί να κάνει μια χώρα μόνη της ε, καλύτερα από ό,τι θα το κάναμε όλοι μαζί. Και νομίζω ότι τώρα το συνειδητοποίησαμε και ακολουθούμε τη σωστή άγουσα. Επίσης, για το ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κοινή εξωτερική πολιτική. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα που ανέφερε προηγουμένως και ο Ρίτσαρτ Χόουιτ. Πριν από δύο μήνες συναντηθήκαμε στο Λονδίνο για τη διάσκεψη του Λονδίνου με θέμα τη Συρία. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κράτη-μέλη ήταν τα δύο τρίτα των υποσχέσεων δωρεών. Και γι' αυτό στέφθηκε με επιτυχία η διάσκεψη του Λονδίνου για τη Συρία. Πέραν του τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε προτείνει ένα οικονομικό σύμφωνο για το Λίβανο και την Ιορδανία με καινοτόμε και δημιουργικές ιδέες το πώς θα γίνει η βιώσιμα μεσοπρόθεσμα το γεγονός ότι η Ιορδανία και το Λίβανο έχουν υποδεχθεί τόσους πολλούς πρόσφυγες και σε καταβλισμούς και σε κοινότητες και πώς ε, θα βοηθήσουμε τις δύο χώρες. Αυτή η ιδέα τώρα δρομολογείται και την αναλύουμε από κοινού. Ακριβώς επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει για την εξυπηρέτηση αυτής της ιδέας και εργαλεία όπως το εμπόριο, ώστε να δημιουργήσουμε αυτό το οικονομικό σύμφωνο ε, για αποφάσεις που είναι αρμόδια να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι κάποιο μεμονωμένο κράτος μέλος. Φαϊνή ήταν η ιδέα του Ηνωμένου Βασιλείου και βοηθά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τους γειτονές και κατέστη δυνατή εφαρμογή της χάρη στην κοινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την εφαρμόσει. Οπότε όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Δεν είναι μόνο win-win κατάσταση, είναι win-win-win για το Ηνωμένο Βασίλειο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις γειτονικέ χώρες. Όλοι βγαίνουν κερδισμένοι, αντί να έχουμε έναν και μόνο χαμένο. Βέβαια έχουμε ακόμη δυσκολίες, έχουμε όρια, έχουμε αδυναμίες, αλλά ο ρόλος μας δεν είναι να πούμε τι δεν λειτουργεί. Εμείς ως ηθήνοντες ε, ε, πολιτικής ε, έχουμε το καθήκον να κάνουμε τα πράγματα να δουλέψουν και να λειτουργήσουν και αυτό προσπαθούμε. Ευχαριστούμε πολύ εδώ.